Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τώρα ε, κοντεύει να τελειώσει η Ολομέλεια, σε ένα-δυο και θα τελειώσει, επομένως καλό είναι να ξεκινήσουμε, γιατί ήδη πέρασε η ώρα. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον ε, ε, ε, ο κύριο Μάρου Σεφκοβίτς, επίτροπο και μελλοντικό αντιπρόεδρο, υποψήφιο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε αυτή την τελευταία ακρόαση για φέτος. Εδώ υπάρχουν τα μέλη δύο επιτροπών, Ήτρα και Ένβη Και μια και βλέπω ότι είναι πολύ οι παριστάμενοι, ε, καλό θα ήταν να κάνουμε φαίνεται τέτοιες κοινέ συνεδριάσεις και εκτός ακροάσεων. Εν πάση περιπτώσει, θα θέλαμε να σας ε, ε, καλωσορίσουμε εδώ. Ε, και να καλωσορίσουμε και τους ε, όσους την παρακολουθούν γιατί είναι μια ανοιχτή ακρόαση. Έχουμε εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, επίσης ε, εκπροσώπους από τη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και μέσω διαδικτύου αυτήν την ακρόαση, μέσω του site του Κοινοβουλίου. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους. Κύριε Σεύκοβιτς. Ήδη ε, είχατε μια ακρόαση ε, ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών ε, για την θέση του Επιτρόπου Μεταφορών και Εμπορίου. Οι δύο επιτροπές ε, απεφάνθησαν ότι ο κύριος Σεύκοβιτς ε, έχει όλα τα προσόντα τα οποία χρειάζονται ε, για να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά στην Κομισιόν. Επομένως, εμείς σήμερα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα νέα ε, χαρτοφυλάκια του ε, Επιτρόπου ε, Σεύκοβιτς όσον αφορά την ενέργεια. Βεβαίως η Επιτροπή μας ασχολείται ιδιαίτερα με την ενέργεια, την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια της ενέργειας, την χρήση, την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς επίσης και την ε, προώθηση της διασύνδεσης των δικτύων ενέργειας. όλα αυτά τα σημεία τα οποία ανέφερα οπωσδήποτε ε, θα αποτελέσουν προτεραιότητες ε, για την επόμενη ε, θητεία και τα μέλη της Επιτροπής μας περιμένουν να δουν τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Εύκοβιτς θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα και, τα, και τις προκλήσεις. Έχετε λάβει ένα έγγραφο εκ των προτέρων συγκεκριμένα το mission letter του ε, κυρίου Σεύκοβιτς, υποψηφίου για τα θέματα ε, ενέργειας. Έχετε λάβει το CV του, το βιογραφικό του, έχετε λάβει επίσης το έγγραφο με, τα, ε, με τη δήλωση συμφερόντων του, καθώς επίσης και το ερωτηματολόγιο στο οποίο έχει απαντήσει. Επίσης η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, Γιούρι, Ε, είχε συνεδρίαση σήμερα στις 6 και δεν έχουμε ακόμα λάβει... Α, το λάβαμε. Λάβαμε την επιστολή και από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ναι, τα, τα, πριν από δύο-τρία λεπτά τη λάβαμε την επιστολή. Και θα την μοιράσουμε την επιστολή αυτή. και αύριο το πρωί θα συζητηθεί στην ε, συνεδρίαση που θα έχουν οι συντονιστές μας, στην ε, συνεδρίαση αξιολόγησης. Ο συμπρόεδρος Λαβία, παρακαλώ, μπορεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Μπούζεκ και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο και ε, υποψήφιο Αντιπρόεδρο για τα θέματα της ενέργειας, τον κύριο Σεύκοβιτς. Ε, γνωρίζουμε την πορεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβακίας, την διπλωματική του πορεία. Το 2004 ήταν ε, ε, μόνιμος αντιπρόσωπος της Σλοβακίας παρά την Ευρωπαϊκή Ενώση. Επίσης ασχολήθηκε με θέματα αθλητισμού, νεότητας και πολιτισμού στην Κομισιόν μέχρι να αναλάβει λάβει το χαρτοφυλάκιο των ε, Διαθεσμικών ε, οργάνων στην Επιτροπή Μπαρόζο 2. Το 2014 το Μάιο εξελέγει ε, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ε, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής ε, ε, Περιβάλλοντος και έχω τη μεγάλη αυτή τιμή και βεβαίως είμαστε ιδιαίτερος, δείχνουμε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα οποία πρόκειται ο πρόεδρος Σεύκοβιτς να αναλάβει. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος περίμενε εδώ και πολύ καιρό αποτελεσματική και φιλόδοξη πολιτική περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη οικονομίας, μιας οικονομίας πράσινης και αηφόρου ε, με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Ο ε, Επίτροπος ε, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης που θα είναι μακρόθωρη από τη μία και αηφόρος από την άλλη. Επομένως χρειαζόμαστε μια κοινή, ενωμένη και ισχυρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν και της των Παρισίων του 2015 εν ώψη όλων των διακυβευμάτων και των μελλοντικών συμφωνιών όπου θα πρέπει να εκπροσωπεί με ισχυρό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ε, να αναπτυχθεί η πράσινη οικονομία και να γίνει η Ευρώπη η ηγέτιδα όσον αφορά την, ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυρίως εν ώψη του ορίζοντα 2030 θα ήθελα να πω και να υπογραμμίσω ότι ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ε, καλή ε, πράσινη οικονομία και να είναι αηφόρα και βιώσιμη θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε ένα νέο σύστημα ανταλλαγής ε, ρήπων. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε, περιμένουμε να ακούσουμε μεγάλη προσοχή αυτά που θα μας πείτε. Ξαναδούν το λόγο σας να Μπούζεκ. Λοιπόν, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο ε, κύριος Εύκοβιτς θα κάνει μία εισαγωγή 13 λεπτών και μετά 5 λεπτά ε, στο τέλος θα ξαναμιλήσει. Μετά την εισαγωγή του ε, κυρίου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είναι ήδη και τώρα Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχουμε χρόνο για 41 ερωτήσεις από τους ε, βουλευτές. Η, η, η ομάδα FDD δεν έχει δώσει ερωτήσεις. Τρία λεπτά θα έχει κάθε ερώτηση. Ένα, δύο λεπτά η ερώτηση, ένα η απάντηση ping-pong σύστημα δηλαδή. Και θα έχουμε τους εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων ε, στην αρχή και τα υπόλοιπα βάσει του, 6, του κανόνα 662. Παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε όλο το χρόνο ομιλίας. Θα έχουμε ανοχή 10 ε, δευτερολέπτων για τον ε, Επίτροπο και 5 για τα μέλη. Μετά από αυτό το όριο ανοχής θα κλείνει το μικρόφωνο δυστυχώς. και πριν από το τέλος του κάθε χρόνου ομιλίας, 10 ε, δευτερόλεπτα, θα αναβοσβήνει ένα φωτάκι. Διερμηνία υπάρχει σε όλες τις γλώσσες, αλλά παρακαλώ πολύ να θυμάστε ότι δεν πρέπει να μιλάτε γρήγορα, γιατί χρειαζόμαστε ε, καλή διερμηνία αποτελεσματική προς 22 χώρες. Κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε υποψήφιε ε, για τη θέση του Αντιπροέδρου, παρακαλώ.